Καθίστε στις θέσεις σας, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη ή μάλλον πριν περάσω εκεί να αναφερθώ στα πρακτικά. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Δεν φαίνεται να υπάρχουν παρατηρήσεις, συνεπώς θεωρούνται δεκτά. Ας περάσουμε στη συζήτηση η οποία προβλέπεται, οι δηλώσεις δηλαδή του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης